So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter mit der Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses und bedanken uns bei den Kollegen. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε λοιπόν την συνεδρίασή μα. Είμαστε τώρα στο σημείο υπαριθμών 8 τη ημερήσια διάταξη προ ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο καλυμμένων ομολόγων. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα, τον κύριο Λούκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδης ηγητές και τους ε, υπόλοιπους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν ε, τροπολογίες στη δική μου την έκθεση. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το κλίμα συνεργασίας που δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ουσιαστική σύγκληση απόψεων στο ότι δεν πρέπει να διαταράξουμε μία εύρυθμα λειτουργούς αγορά και δεν επιθυμούμε να επιφέρουμε καμία αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση, οποτεδήποτε μιλάμε για καλυμμένα ομόλογα. Άρα δηλαδή η δική μου έκθεση τι λέει, λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει να απαγορεύσουμε προϊόντα στην αγορά, αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να θέσουμε τις ε, συνθήκες πλαίσιο που θα διευκρινίζουν ε, ποια ε, προϊόντα δικαιολογούνται έτσι ώστε να είναι και ρυθμιστικά προτιμητέα, ας το πούμε. Αυτά δηλαδή που αφορούν στα καλυμμένα ομόλογα. Αυτό είναι το πνεύμα της έκθεσης και προς αυτή την κατεύθυνση ε, τίνουν και αρκετές τροπολογίες. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι υπάρχει ουσιαστική συμφωνία στο ότι δεν θα πρέπει να επέμβουμε σε αυτά τα καλυμμένα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ήδη στο παρελθόν. Μιλάμε για κάτι το καινούριο, για καινούρια καλυμμένα ομόλογα τα οποία ε, θα φορούν στο μέλλον. Σας επαναλαμβάνω, όχι εκείνα τα οποία ήδη βρίσκονται στην αγορά. Βλέποντας λοιπόν τις ε, τροπολογίες, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν τρία θέματα ε, όπου θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Τρία θέματα τα οποία βέβαια αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Καταρχήν αφορά το διαχωρισμό ε, ανάμεσα στα καλυμμένα ομόλογα, αφενός αυτό όπως τα γνωρίζουμε, με την μεγαλύτερη κανονιστική προτίμηση. Έτσι θα τα χαρακτηρίζαμε. Αυτό αφενός και αφετέρου αυτά ε, από την άλλη είναι ε, τα εργαλεία εκείνα, ένα διαφορετικό χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο εμείς ε, το παρουσιάζουμε ως καλυμμένο ομόλογο και αυτό θα μπορούσαν, αυτά θα μπορούσαν να είναι προτιμητέα από τις τράπεζες και από τους χρηματοψηφιακούς οργανισμούς, όμως αυτά δεν δίνουμε την ύψιστη προτίμηση. Υπάρχουν κατά τα άλλα και άλλες απόψεις, διστάμενες απόψεις. Το πώς δηλαδή ορίζουμε τα καλυμμένα ομόλογα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επιτρεπόμενες περιουσιακές κατηγορίες. Όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τιτλοποιήσεις και σε κρατικά ομόλογα. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις και από την άλλη μοιάζει να συμφωνούν όλοι ότι τα δάνεια για τις υποδομές και τα δάνεια για ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι καλυμμένα ομόλογα. Θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε και για θέματα ανταγωνισμού. Θα ήθελα εδώ να αφαιρθώ κυρίως στο τι θα κάνουμε με κινητές αξίες όπως είναι τα σκάφη. Υπάρχουν άλλα ε, αντικείμενα όπως τα αεροσκάφη. Αυτά δεν προτιμούνται, ούτε και τα τρένα υψηλή ταχύτητας. Εγώ θεωρώ ότι εδώ όμω υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού προς όφελος των σκαφών και μόνον αυτό, αλλά τα καλυμμένα ομόλογα ε, όταν είναι σε σκάφη είναι ομόλογα που έχουν σχέση με ε, κρατικά ομόλογα ή ενυπόθηκα δάνεια. Και αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Το δεύτερο πολύ σημαντικό που θέλω να σας δείξω αφορά την παράταση της διάρκειας ισχύως. Δηλαδή αυτό που λέγεται soft bullets και conditional pass through. Αυτές είναι δύο, δύο εργαλεία τα οποία αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην αγορά. Εγώ λέω τα soft bullets να τα αφήσουμε, να τα επιτρέψουμε για ένα χρόνο όμως. Και στα soft bullets εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει αυθαίρετη εφαρμογή του εκδότη. Αλλά όσον αφορά τα εργαλεία και τη χρήση αυτής της ε, δομής των soft bullets θα πρέπει να υπάρχει και η συγκατάθεση της εποπτικής αρχής. Και από αυτού υπάρχει η διάσταση απόψεων. Μερικοί πιστεύουν ότι τα soft bullets θα πρέπει να είναι συνάρτηση κάποιων μακροοικονομικών συνθήκων. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να οριστεί, γιατί θα πρέπει να ορίσουμε ποιες ακριβώς μακροοικονομικές συνθήκες είναι αποδεκτές και ποιες όχι. Αυτό όμως δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Και μόνο αυτό, αλλά θεωρώ ότι και ο κίνδυνος του εκδότη, το να μετακυλείται αυτό στον επενδυτή, νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει συστημικές αντιδράσεις, τις οποίες και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε. Τρίτο θέμα τώρα και με αυτό θα κλείσω έχει σχέση με τις μεθόδους αξιολόγησης. Επ' αυτού έχουν κατατεθεί κάποιες τροπολογίες και νομίζω εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις ονομαστικές αξίες ε, γιατί υπάρχουν κάποια ομόλογα τα οποία ε, σαφώς ε, και είναι κάτω από την ονομαστική αξία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με την έννοια ότι αν η αγορά είναι ανωδική για τις ονομαστικές αξίες, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Να ληφθεί υπόψη για να μειωθούν τα collaterals, οι εγγύησεις. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα τους σκιώδες εισηγητές Τάριου Σολοζάτη για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον κύριο Λουκέ ε, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Νομίζω ότι η ιδέα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα είναι καλή. Πρόκειται για μια αγορά η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και σίγουρα δεδομένου ότι υφίστανται μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών και κανονισμών χρειάζεται να γίνει μια προσπάθεια ώστε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο να καταστεί πιο αποτελεσματικό και σταθερό. Τώρα, δεχόμενη τη γενική αυτή ιδέα εργασίας, ε, ε, θα έλεγα ότι θα ήταν μάλλον προώρο να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες αυτού του πλαισίου, διότι μας λείπουν βασικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς και τις πιθανές την πιθανή, τις πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών που θέλουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε κάποια μελέτη επιπτώσεων για την αγορά καλυμμένων ομολόγων στην Ευρώπη και για το πώς ε, οι προτινόμενες αλλαγές θα επηρεάσουν συγκεκριμένους τομείς αυτής της αγοράς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ίσως να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτού του θέματος, να βελτιώσουμε τη συνεργασία με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία και τεκμήρια που θα μας ε, δώσουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε το πώς θα επηρεαστεί η αγορά και οι εργασίες της από έναν πιθανό κανονισμό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ε, χαιρετήσω αυτή την ε, προσέγγιση που βασίζεται σε αρχές και δεν επιζητά μια εναρμόνιση σε, όλο το, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παρά μόνο μέσω ε, ε, εθνικών λύσεων. Να μην έχουμε συγκεκριμένους κανόνες λοιπόν. Θα πρέπει να πω ότι σε πολλές εθνικές αγορές για τα καλυμμένα ομόλογα υπάρχουν περιπτώσεις εφαρμογής διαφορετικών λύσεων και οι τομείς των καλυμμένων ομολόγων λειτουργήσαν πολύ καλά για πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν, εφόσον λειτουργεί καλά το πράγμα, δεν υπάρχει άμεσος λόγος να αλλάξουμε την κατάσταση, ε, ε, εκτός αν υπάρχει όντως λόγος και αποδείξουμε ότι οι ε, αλλαγές που θα επιφέρουμε θα κάνουν την κατάσταση ακόμα καλύτερη. Αυτά είναι τα γενικά μου σχόλια. Τώρα θα έλθω στα τρία σημεία που ανέφερε ο εισηγητής. Πρώτον, ορισμός των καλυμμένων ομολόγων προς το παρόν δεν έχουμε ξεκάθαρο ορισμό. Αυτό ισχύει. Υπάρχει μια ε, πρακτική ε, που ε, χρησιμοποιεί την οδηγία ως ΕΚΑ ως σημείο έναρξης. Ε, δηλαδή, ο κύριος Λίκε είπε ότι θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα ομόλογα που ε, συμμορφώνονται με το άρθρο 1 προς 9 του CRR, του Κανονισμού για τις Κεφαλαϊκές απαιτήσει. Ως προς την έκδοση λοιπόν των καλυμμένων ομολόγων, ε, στην ουσία εξαιρείται μια κατηγορία καλυμμένων ομολόγων που εκδόθηκαν στο παρελθόν και είναι διαφορετικές από αυτές που ε, αναφέρονται στο άρθρο 129. Συμφωνώ με τον κύριο και επίσης ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα κινδύνου που σχετίζονται με τις διάφορες κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού. Για παράδειγμα, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι ε, σε ίση μοίρα τα καλυμμένα ε, ομόλογα που έχουν εξασφάλιση από το κράτος με αυτά που καλύπτονται μέσα από ε, πλοία, για παράδειγμα. Διότι τα πλοία δεν είναι το ίδιο αξιόπιστα με τα ενυπόθηκα δάνεια ή το δημόσιο χρέος. Αυτά τα έχουμε ήδη συζητήσει. Φυσικά, εκτός από τα πλοία υπάρχουν και άλλα ε, στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα ε, τα ενυπόθηκα δάνεια ή τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εις δείτε, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Αυτοί οι τομείς της αγοράς έχουν λειτουργήσει πολύ καλά ως τώρα και θεωρώ ότι δεν πρέπει να καταστρέψουμε κάτι που έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποδοτικά, ε, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και τον παράγοντα του κινδύνου. Αυτό που προτείνει ο κύριος Λουκέ ε, είναι καλυμμένα ομόλογα premium κατηγορίας ε, που ε, συμμορφώνται με τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσει, αφαιρώντας βέβαια τα πλοία και θα δούμε τώρα ποια θα είναι τα καλυμμένα ομόλογα τα οποία θα είναι στην κατηγορία των European Secured Notes, η νέα κατηγορία που προτείνεται. Εγώ θα πρότεινα τρεις κατηγορίες καλυμμένων ομολόγων. Η πρώτη θα ήταν τα premium καλυμμένα ομόλογα που πρότεινε ο κύριος Λίκε. Η τρίτη, ε, αυτά που υφίστανται ήδη και εφαρμόζονται στην πράξη ε, και όλα τα άλλα που δεν συμμορφώνονται θα είναι τα λεγόμενα European Secured Notes. Τώρα, δύο λόγια ε, για τα, την ε, παράταση στην ημερομηνία λήξης και θα τελειώσω. Δεν ξέρω αν αυτό περνάει τον κίνδυνο από τους ασφαλιστές, τους επενδυτές. Νομίζω ότι οι επενδυτές έχουν αρκετό περιθώριο να επανακάμψουν και αν θέλετε να το συζητήσουμε. Εγώ θα ήμουν υπέρ μεγαλύτερων παρατάσεων για τις μεθόδους τώρα αξιολόγησης όταν αξιολογούμε την ε, αξία των ε, στοιχείων του ενεργητικού. Ε, η κάθε χώρα έχει τη δική της νομοθεσία και τη δική της πρακτική. Ας το αφήσουμε σε αυτούς λοιπόν. Ευχαριστώ. Επειδή ούτως ή άλλως έχουμε χάσει χρόνο, είμαστε πίσω επειδή η προηγούμενη ε, συνεδρίαση πήρε περισσότερο χρόνο, θα είναι σημαντικό να είμαστε πιστοί στο χρόνο. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Πάμε λοιπόν στον ε, Άλφρεντ Σάντα από το S&D. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, προσέγγιση του, την επικοδομητική, στην προσπάθεια να βρεθεί ένα συμβιβασμό στο πλαίσιο του κειμένου αυτού. Όλοι συμφωνούμε ότι μια πιο, ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές. Τα εθνικά σύστημα, συστήματα έως τώρα έχουν λειτουργήσει πολύ καλά και δεν πρέπει να ε, παρεμποδιστεί η λειτουργία τους. Θέλω λοιπόν να έχουμε μια ελαφριά προσέγγιση στην νομοθεσία αυτή, να βασιστούμε σε αυτά που έχουν γίνει έως τώρα. Ο κλάδος έχει αποδώσει σωστά και δεν πρέπει να περιορίσουμε την αγορά με νέους κανόνες και πηγαίνοντας πέρα ε, από αυτά που έχει πετύχει η ίδια η αγορά. Ο βασικός συμβασμός είναι ο εξής. Ό,τι έχει λειτουργήσει καλά δεν πρέπει να παρεμβολιστεί στη λειτουργία του. Αν δούμε τις εθνικές πρακτικές, ε, δεν πρέπει να περιορίσουμε τις εθνικές πρακτικές, διότι έως τώρα έχουν στεφθεί από επιτυχία. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, Δύο έχω υποβάλει εγώ με βάση ζητήματα που έχουν συζητηθεί ήδη ο ορισμός αυτών των ε, και καλυμμένων ομολόγων, ομολόγων. Πρέπει όλα, αυ, όλα αυτά τα ομόλογα να είναι οσεκά. Επίσης αυτά που συμμορφώνονται με το CRR δεν πρέπει να έχουν προτιμησιακές συνθήκες κινδύνου. και δεν πρέπει βεβαίως να υποβαθμίζονται σε ESN. Δεν θα συνδέσω τον ορισμό των κεκαλυμμένων ε, ομολόγων με τους ορισμούς όπως λέει ο μιλητής διότι αυτό περιπλέκει το σύστημα. Αν υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι φορά τις κεφαλαϊκές ε, θα βρεθούμε πιο δυσκολιών. Η Κομισιόν μόλις δημοσίευσε μια μελέτη που πάει προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε. Θα πρέπει να ε, ορίζεται ως οσεκά δηλαδή το καλυμμένο ομόλογο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπόκεινται στους ίδιους κανόνες. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα δάνεια υποδομών ε, γνωρίζω ότι ο συγκριτής δυσκολεύεται με αυτό, θεωρεί ότι δεν πρέπει να καλύπτονται, ε, να εμπίπτουν σε καλυμμένα ομόλογα, αν και ορισμένε φορέ οι ίδιε πρακτικέ χρησιμοποιούνται. Θεωρώ ότι έχει δίκιο ο συγκριτής, αλλά ας αφήσουμε τον νομοθέτη, τον εθνικό, να πάρει την απόφαση ε, αναπερίπτωση. Με βάση αυτά που προτείνονται, μπορούμε να αναφερθούμε στην ανησυχία αυτή που υπάρχει, αλλά ας αφήσουμε ένα περιθώριο λιγμών σε εθνικό επίπεδο. Δεν ξέρω αν θα αρέσει τον εισηγητή αυτό. Τώρα για την οριμότητα. Βεβαίω δεν πρέπει, να, δεν πρέπει να υπάρχει επέκταση επάπειρων. Η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Ισπανία είναι οι μόνες χώρες που ισχύει κάτι άλλο, αλλά και εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Σε όλες τις άλλες δικαιοδοσίες Ακολουθείτε αυτή η οδός. Υπάρχει δηλαδή επέκταση ε, σε ό,τι αφορά την οριμότητα, αλλά υπό πολύ συγκεκριμένε προποθέσει. Και κάτι άλλο για την υπόθηκα δάνεια στη Γαλλία. Μια τροπολογία αποκλείει αυτά τα δάνεια, διότι δεν είναι εν υπόθηκα δάνεια ακριβώς. Είναι ε, δάνεια διαμονής αλλά είναι 40% της αγοράς στη Γαλλία. Έως τώρα έχει λειτουργήσει καλά το σύστημα. Γιατί είναι στεγαστικά δάνεια. Κάτι που λειτουργεί σωστά πρέπει να συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε. Είναι μια ιδιαιτερότητα της γαλλικής αγοράς και δεν νομίζω να πρέπει να προσπαθούμε εμείς να μαντέψουμε τι είναι καλό για την αγορά. Όταν έχουν λειτουργήσει καλά τα πράγματα πρέπει να το στηρίξουμε. Βεβαίως εισηγητής ε, λέει μενα πολύ καλά πράγματα σε σχέση με το, τα assets, τα στοιχεία που θα πρέπει να μπορούν να, να συμπεριληφθούν εδώ στο στοιχείο ενεργητικού δεν έχει υπάρξει και πάλι κανένα πρόβλημα έως τώρα. Γιατί να μιλήσουμε λοιπόν για τα back CBs εδώ Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ για του φιλελεύθερου η κόρα, αλλά νομίζω η κυρία Βίρινγκ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της Κόρα που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ γιατί είχε αναλάβει άλλες υποχρώσεις. Η Κόρα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης και για τις συμβαστικές προτάσεις που κατέθεσε και που έλαβε υπόψη κάποιες τροπολογίες δικές της. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε ότι τα καλυμμένα ομόλογα, η αγορά τους αυτή τη στιγμή λειτουργεί πολύ καλά στην Ευρώπη και τα εθνικά πλαίσια για τα προϊόντα αυτά ήδη υπάρχουν. Στην Ολλανδία ε, τέθησε σε ισχύ το 2015 πλήρης αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τα καλυμμένα ομόλογα. Πρέπει βέβαια να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα που θα βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές που θα ορίσει η τράπεζα, η υποπτική αρχή τραπεζών στη δική της την έκθεση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή που εξέδωσε το 2014. Όπως προτείνει λοιπόν η εποπτική αυτή αρχή, θα πρέπει να ισχύουν προδιαγραφές υψηλής ποιότητας και βέλτιες πρακτικές της αγοράς, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το εκάστοτε εθνικό καθεστώς, χωρίς να διαταράσετε το εθνικό σύστημα. Η ιδιαιτερότητα των εθνικών νομολογιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και παράλληλα να υπάρχει αρκετό περιθώριο ευελιξίας. Επίσης, να υπάρχει ε, η προσπάθεια αποφυγή υπερβολικού διοικητικού άχθους. Όσον αφορά τώρα την ιδέα του να υπάρχουν ευρωπαϊκά καλυμμένα ομόλογα, αυτό που προτείνει ο συγητής, ε, η σκιώδη συγήτρια της ε, των Φιλελευθέρων ε, διερωτάται κατά πόσον θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Κομισιόν να μας εξηγήσει τη δική στην άποψη και αυτό θα μας βοηθούσε στο να καταλήξουμε κατά πόσον το ESN επιτρέπει τη διαφοροποίηση των προϊόντων και παράλληλα παράλληλα το να μην υπάρξει ζημιά που να προκληθεί στην παραδοσιακή αγορά των ε, καλυμμένων ομολόγων. Η σκιώδη συγκήτρια των Φιλευτέρων προσβλέπει στη συζήτηση επί του θέματος με στόχο να επιτευχθεί ε, κοινή στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ ωραία. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ε, πάρα πολύ σύντομα θα σας πω αυτό που θέλω να πω, χωρίς να επαναλάβω αυτά που ελέγξαν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, να σας πούμε ότι παρακολουθούμε αυτό τον επικοδομητικό τρόπο προσέγγισης όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα. Κοιτάξτε, αυτά που λειτουργούν καλά πρέπει να τα διατηρούμε και γι' αυτό το λόγο εμείς στηρίζουμε αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Έχουμε βέβαια κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά τη δημιουργία ενός νέου τίτλου του ESN. Ε, εδώ έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την κατουσία. Πρόκειται για ένα υβριδικό εργαλείο αν δούμε τις σχετικές ε, προτάσεις ε, και αν δούμε το τι ισχύει για τις τιτλοποιήσεις και για τα καλυμμένα ομόλογα μέχρι τώρα, κατ' ουσίαν πρέπει να πρόκειται. Πρόκειται για εξασφάλιση με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η αγορά θα μπορούσε αυτό να το εκλάβει ως μία εξασφάλιση που όμως ε, αυτή η εξασφάλιση τελικά μπορεί και να μην συμβαδίζει με την πραγματική αξία του προϊόντος. Εγώ νομίζω ότι μόνο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ως ε, δική μας διαφορετική άποψη. Πάντως μας ενδιαφέρει να παρακολουθήσουμε την όλη αυτή δουλειά και με την ε, κατάθεση τροπολογιών, γιατί αν αυτό το ε, προϊόν, το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα συμβιβασμού, να παραμείνουν τα καλυμμένα ομόλογα όσοι έχουν τώρα. Αυτή είναι μια κάποια λίστα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνούμε όλοι από αυτού. Ο κύριος Βεν Γκίγκολτ εκ μέρους των Πρασίνων. Εκτός μικροφώνου. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την καλή συνεργασία και τον εισηγητή. Εμείς με την κατευθυντήρια γραμμή που έχει προτιμηθεί συμφωνούμε. Ως τώρα ε, λειτουργεί πολύ καλά αυτή η αγορά. Στην ουσία, εμείς λοιπόν πρέπει από την ευρωπαϊκή πλευρά να προσέξουμε ώστε να μην έχουμε περισσότερη ζημιά παρά ωφέλη. Απ' την άλλη, είναι πολύ σημαντικό στον τομέα των καλυμμένων ομολόγων να βοηθήσουμε την κεφαλαία αγορά και γι' αυτό χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα γι' αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια θετική ανοιχτή πρόσβαση. Αυτό φαίνεται μέσα από την έκθεση και πέρα από αυτό, από ό,τι φαίνεται, αν ε, συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να προσέχουμε τα στάνταρ να είναι ε, υψηλά Ε, επιπλέον υπάρχουν κάποια στοιχεία, κάποιες λεπτομέρειες που παραμένουν ανοιχτά θέματα. Το γεγονός που ανέφερε ο εισηγητής, ε, τα κριτήρια ε, προτίμησης στον κανονισμό για τις κεβαλαϊκές απαιτήσει, μιλάμε για τα πλοία τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μια ένα προτιμησιακό καθεστώς σε σχέση με άλλους τομείς που είναι ιδιαίτερα ασφαλείς. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέξεις, αυτό χαιρόμαστε που υφίσταται, όμως σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό ε, να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτό θα στρέβλωνε την αγορά. Και η πρόταση του Άλντε, ε, το να έχουμε ένα impact assessment, είναι ένας λογικός δρόμος να ακολουθήσουμε. Επίσης, η αποτίμηση των τιμών αγοράς είναι κάτι που ως τώρα υπάρχει ως πρακτική, όμως οδηγεί σε μεγαλύτερη ανασφάλεια, πολύ γραφειοκρατία, γίνεται πιο ακριβό το προϊόν, το οποίο ως τώρα ήταν σχετικά απλό και λειτουργούσε καλά. Πολλές φορές κανείς ε, θα μπορούσε να υποθέσει ότι θα είχαμε διαφορετικές τιμές ε, στα κρατικά ομόλογα και ειλικρινά νομίζω ότι θα έπρεπε να αποφύγουμε μια τέτοια μορφή αποτίμησης. Δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και κατά τα άλλα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φωνστόλ δεν είναι εδώ για το EFTD, ο κύριος Άνεμανς για το ΕΝΕΦ. Να πω γεια στον συνάδελφο Λούκη και θα μιλήσω Ολλανδικά. Όταν κοίταξα το σχέδιο της έκθεσής σας, δεν ε, είδα ουσιαστικά κάτι συγκεκριμένο για τα καλυμμένα ομόλογα. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να υποστηρίξω την πρότασή σας για τον ορισμό, για τη διαφάνεια. Θα προτιμούσαμε μία άλλη λύση, αλλά υπάρχουν και δύο τροπολογίες στο συμβασμό που μόλις είδαμε, οι οποίες φαίνεται ότι οδηγούν σε παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στα πλαίσια της ε, Ένωσης ε, των, της, των κεφαλαγορών, της αγοράς κεφαλαίων. Ο συμβιβασμός ε, για τον ορισμό στην ουσία θα δημιουργήσει προβλήματα με την εθνική νομοθεσία και τον ορισμό. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις που πάνε πέρα από την προηγούμενη έκθεση. Το σχέδιο της έκθεσης ήταν αποδεκτό για εμάς. Τώρα με τις τροπολογίες νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Οπότε φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Περάμε τώρα στο Catch the Eye. Ένα λεπτό όμως πραγματικά, διότι θέλει ε, να μιλήσει ε, και ο εισηγητής και κανονικά είχαμε διαμείνει μέχρι τις 12 μόνο. Η κυρία Μπερές, ευχαριστώ πρόεδρε, πολλά υπόθηκαν. Εγώ θέλω να επανέλθω σε τρία σημεία δεν μπορούμε να ξεκινάμε με το δεδομένο ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την αγορά εκεί όπου λειτουργεί σωστά ε, και οι εθνικές πρακτικές ε, που δεν είναι ε, ίδιες με αυτές τις χώρες από την οποία πρέπει το εισηγητής να αναλλάξουν, έτσι. Το είπε ο κύριος Σαντ από τους, από τους σοσιαλιστές, το, το είπε και το ΕΛΚ. Πιστεύω το θέμα της χρηματοδότησης για τις εγγυήσεις ε, ε, σε τέτοια είδους δάνεια πρέπει να παραμείνουν. Διότι ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα. Ήταν ένας καλός τρόπος χρηματοδότηση. Ε, το δεύτερο, σε σχέση με το χρέος, δεν πρέπει μέσω αυτών των πρακτικών η χρηματοδότηση του χρέους των κρατών να περιπλακεί ακόμα περισσότερο. Και τρίτον, Συμφωνώ με τον Σβέν Ίγκολ. Αν πρέπει να περάσουμε δηλαδή από μια ονομαστική αξία σε μια αξία αγοράς. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ που χρειάζεται αξιολόγηση αντικτύπου όταν γνωρίζουμε την πλητικότητα των αγορών. Είπε ο εισηγητή ε, ότι αυτό θα είχε νόημα, ότι είναι λογικό να γίνει αυτό όταν έχουμε ε, άνοδο, αλλά όταν έχουμε πτώση δεν μα είπε τι θα συμβεί. Μια αλλαγή λοιπόν τη τιμή αναφορά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην περίπτωση αυτή. Μάλιστα, θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Λιντιέ Μιλογό έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί καλωσορίζουμε το σχέδιο ε, έκθεσης του Ευρωπαϊκού στα πλαίσια της συζήτησης που γίνεται για τα κεκαλυμμένα ομόλογα, ε, που πρέπει να παραμείνει ένας, ε, μια πηγή χρηματοδότηση αποτελεσματική στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία με την αρμόνιση σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια στο προαπαιτούμενο ότι αυτό δεν πρέπει να διακυβεύει τα εθνικά μοντέλα και την λειτουργία του, τη λειτουργικότητά του. Στη μελέτη η οποία δημοσιεύσαμε φτάνει στο συμπέρασμα ότι τα ωφέλη από έναν αρμονισμένο πλαίσιο είναι πολύ μεγαλύτερα από το κόστο. Η Κομισιόν λοιπόν εξετάζει τώρα τη δυνατότητα ε, να πάει προ μια εναρμόνιση που βασίζεται στι αρχέ, να βασίζεται σε αυτά που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο, όπω άλλωστε αναφέρει και η έκθεση EPA. Ε, βεβαίως στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης για την Κεφαλιακή Ένωση θα εξεταστεί και αυτό. Οποιοδήποτε, ένα, ένα σημείο κλειδί είναι η, η σύγκληση των καλυμμένων ομολόγων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ε, τάξεις. Αυτά ε, τα οποία υπόκεινται σε ΟΣΕΚΑ και αυτά που υπόκεινται στο CRR. Αυτό δημιουργεί μια στέρεα δομή μας επιτρέπει να επιλύσουμε τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν για τα πιο ασφαλή ομόλογα ε, καλυμμένων ομολόγων παρότι δεν είναι ίδιες οι απαιτήσει, υπάρχει μια κάποια αναγνώριση ως και καλυμμένο ομόλογο και για τα άλλα ομόλογα. Θεωρείται ένα μια ασφαλής επένδυση για τα usage, θεωρείται ένα ε, όργανο διαχείρισης ρευστότητας για τις τράπεζες. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει το σύστημα αυτό με τέτοιο τρόπο που να ε, δυσκολεύει τη λειτουργία του. Ε, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε Urban Secure Nodes που έρχεται να ε, ε, καλύψει το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια αναφορά επίσης στην αγορά, στο θέμα των CPTs και των soft bullets. Αυτές οι δομές προέρχονται από την αγορά ως πρωτοβουλίες. Και βεβαίω μπαίνουν ζητήματα ρευστότητα, επαναχρηματοδότησης για να αντιμετωπιστεί παραδείγματο χάρη μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά. Εφόσον δεν ρυθμίζονται αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, αλλά χρησιμοποιούνται ευρέω, σημαντικό θα ήταν κατά τη γνώμη μα να πλαισιώσουμε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο τη χρήση αυτών των δομών στα πλαίσια ενό ισχυρού πλαισίου και καλυμμένων ομολόγων. Τελειώνοντα, Πρόεδρε, να πω ότι εμεί καλωσορίζουμε το σχέδιο έκθεση του Ευρωπαϊκή Κοινοβουλία και τη σημερινή συζήτηση. Είναι κάτι που θα ε, εξεταστεί στα πλαίσια τη αποφάση που θα πάρουμε για το αν θα προχωρήσουμε με, νομοθετική διαδικα... με νομοθεσία. Αν προχωρήσουμε με νομοθεσία, θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσω... προσεκτικά, έτσι ώστε ε, να μην διαταραχθεί αυτή η σημαντική πηγή χρηματοδότηση για τι τράπεζε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Και τέλο, ο εισηγητή. Παρακαλώ. Θα μιλήσω λοιπόν ε, τώρα αγγλικά όπως έκαναν και όλοι οι άλλοι. Να ευχαριστήσω όλους ε, όσοι συνέβαλαν στη συζήτηση για τις ε, παρατηρήσεις τους. Τους ευχαριστώ για τις προτάσεις τους και θα ήθελα να σχολιάσω σύντομα κάποια θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Ροζάτη πρότεινε μία προσέγγιση τρία επίπεδα όσον αφορά τα καλυμμένα ομόλογα. Ε, νομίζω ότι πράγματι αυτό είναι ένας καλός τρόπος για να επιτύχουμε συμβιβασμό. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έχουμε ήδη δύο επίπεδα ε, που έχουν όμως το, το ίδιο όνομα. Μιλάμε για καλυμμένα ομόλογα και δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός σε αυτά τα δύο επίπεδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Άρα δηλαδή πρέπει και νομίζω ότι αυτό που είπατε καλή προσέγγιση. Ε, όσον αφορά ε, στο, στον κανονισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, εγώ αναφέρθηκα στα σκάφη και είπα ότι εντάξει, ίσως πρέπει να τα αποσύρουμε από την προτιμησιακή τους μεταχείριση μέχρι τώρα, γιατί πράγματι ε, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα επιχειρήματα επ' αυτού. Ε, όσον αφορά το θέμα της Γαλλίας, πράγματι επ' αυτού έχω και εγώ ε, καταβάλει κάποια τροπολογία. εκτιμώ τις ε, εγγυήσεις ε, αλλά θα πρέπει να δούμε λιγάκι και τη σύσταση της ε, εποπτικής αρχής των τραπεζών. Δηλαδή να μπορούν σε αυτές τις εγγυήσεις να προσθεθούν και υπόθεκα δάνεια σε περίπτωση πτώχευσης του χαρτοφυλακίου εξασφαλίσεων. Νομίζω ότι αυτό ε, σωστά το προτείνει η υποπτική Αρχή ε, και εγώ ε, πράγματι θεωρώ ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε αυτές τις εξασφαλίσεις από τον κανονισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η, υπερβολική, μάλλον, η παράταση της οριμότητας τίθεται, τα soft bullets υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό. νομίζω ότι το να πει κανεί μέχρι τώρα τα πήγανε πάρα πολύ καλά γιατί να πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε κάτι, ε, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το 2007 μπορεί να έλεγε κανείς ε, επειδή και οι εξασφαλίσεις ε, πήγαν μια χαρά να μην αλλάξουμε τίποτα. Αυτό μας δεν γίνεται. Μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τους συστημικούς κινδύνους στη νομοθεσία μας. Και όπως είπα ήδη στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις, αυτό που θέλω να κάνω εγώ στην έκθεση είναι να ορίσω με απόλυτη σαφήνεια ποια καλυμμένα ομόλογα ποια, ε, χρέη, ποια εργαλεία του χρέους χρήζουν και μπορούν να έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Αυτό πρέπει να το ρίσουμε με σαφήνεια. Αν είναι καλό ε, να ε, παραταθεί η οριμότητά τους και αυτό να είναι άμεση συνάρτηση μακροοικονομικών εξελίξεων, αυτό πράγματι έχετε δίκιο, θα πρέπει να το συζητήσουμε στη συνεδρίαση των σκιωδών. Εμένα με απασχολεί η συστημική οριμότητα. Επιπτώσεις ε, αντικτύπου, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους και από τον κύριο Σάτη, Αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξετάσουμε κάποια θέματα τα οποία είναι επίμαχα. Ε, αυτή η έκθεση δεν είναι νομοθετική, είναι μήνυ έκθεση. Κατόπιν τούτου δεν ορίζουμε συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να νομοθετηθούν, απλώς δημιουργούμε κάποιο προβληματισμό, εξετάζουμε κάποια θέματα που υπάρχουν και προφανώς και μπορούμε να ζητήσουμε μελέτη αντικτύπου, αλλά απ' την άλλη δεν βλέπω και να υπάρχει πίεση χρόνου για να κατατεθεί συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι κάποιες εξελίξεις στην αγορά ίσως είναι προβληματικές στη στιγμή στιγμή μάλιστα που μεταβάλλεται η αγορά. Και η τελευταία μου παρατήρηση σχετικά με τα ESN θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζω κατ' ουσίαν είναι μια ευκαιρία για τους επιχειρηματίες να μπορούν να χρηματοδοτούν επενδυτικά προγράμματα τη στιγμή που τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες θεσμικές ρυθμίσεις οι οποίες ωφέλησαν όμως άλλου είδους προγράμματα παραδείγματο χάρη τη διπλή προσφυγή ή την ε, δημόσια εποπτεία. Αυτά, ε, μάλλον το να υπάρχει εδώ ε, σύνδεση με την τυπλοποίηση, αυτό μπορεί να αποτελεί μειονέκτημα. Σας λέω, θα μπορούσε να υπήρχε δυνατότητα ε, να καταφύγουν επενδυτές σε θεσμικά εργαλεία που αποδείχθηκαν χρήσιμα και γιατί να, πρέπει να τους στερήσουμε αυτήν την ευκαιρία. Αυτά είχα να σας πω. Εντάξει, ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Τα υπόλοιπα στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Πράγματι, να τα πείτε τα υπόλοιπα, Τα απόγευμα. Φτάνει, η διερμηνή φτάνει μέχρι τώρα. Η ψηφοφορία θα είναι στις 19 Ιουνίου. Ε, μετά στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Επόμενη συνεδρίαση 5η, 8 Ιουνίου. Γεια σας.